Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα σας. Σίγουρα πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλα τα μέλη της Επιτροπής που κατάφεραν να έρθουν σήμερα μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή νύχτα που περάσαμε. Δύο μέρες θα καλύψει η συνεδρίαση της ε, υποεπιτροπής μας Άμυνας και Ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η συνεδρίασή μας και δίδεται προτεραιότητα στη διερμηνία στις γλώσσες των πλήρων μελών της υποεπιτροπής μας, της υποεπιτροπής αυτής Άμυνας και Ασφάλειας. Θα ήθελα ευθύ αμέσω να περάσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουν γίνει κάποιες ε, μικρές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. για την προετοιμασία τη αποστολή αυτή, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή για την εξαιρετική του συμβολή. Θεωρώ ότι ήταν πολύ επικοδομητική η επίσκεψή μα στη χώρα αυτή και θα προβλεφθεί και ένα ειδικό σημείο τη ημερήσια διάταξη για το ζήτημα αυτό και θα καλέσουμε βέβαια και εκπροσώπους και από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το ζήτημα αυτό. Ήθελα να κάνω απλώ μια σύντομη ανακοίνωση για την αποστολή αυτή, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω επί του παρόντος όλους όσοι συμμετείχαν στην αποστολή αυτή και όσοι βοήθησαν στην διοργάνωση της αποστολής αυτής. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί πραγματικά τα πρότυπα ασφαλείας τα οποία παρήχει η Ουκρανική πλευρά ήταν ιδιαίτερα υψηλά Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο ουσιαστικό σημείο της σημερινής μας πρωινής συνεδρίασης. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της δημόσιας αυτής ακρόασης για το Αφγανιστάν, το μέλλον της αποστολής EUPOL, της αστυνομικής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα το πρωί. Αναφέρομαι στον κύριο Μπέρτ Βέρσμεσεν, ο οποίος είναι αναπληρωτής διοικητής της μη στρατιωτικής επιχείρησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Οξτερικής Δράσης και να καλωσορίσω επίσης και τον καθηγητή Έντουαρτ Μπέρκ από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth στον Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ε, ειδικεύεται σε ζητήματα στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, όπως σας είπα. θα μας δοθεί σίγουρα μια πολύ θετική δυνατότητα να μιλήσουμε για τα ζητήματα ασφάλειας στο Αφγανιστάν και στη γύρω περιοχή και θα μας απασχολήσει βέβαια και το γενικότερο μέλλον της αποστολής Ιγιουπόλα. Θα θυμάστε ότι η κυρία Πία Στίεβεν, η επικεφαλής της αποστολής αυτής, είχε έρθει και μας είχε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες και σας είχαμε τότε υποσχεθεί ότι θα δίναμε συνέχεια στο ζήτημα αυτό και ότι θα προβλέπαμε περισσότερο χρόνο για να γίνει μια διεξοδική συζήτηση προτού ληφθεί μια τελική απόφαση τελικά για το μέλλον της αποστολής EUPOL. Σας προτείνω λοιπόν να περάσουμε ευθύς αμέσω στην δημόσια αυτή μας ακρόαση και θα δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Βέρσμεσεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σε ενημερώσω για την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Μπέρκα, θα σας αντικαθιστώ εδώ πέρα τον διοικητή της μη στρατοτική επιχείρησης, ο οποίος σας μίλησε όμως τον Ιούνιο σε μια συνεδρίαση που είχατε αφιερώσει τότε στην αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για τα επιτεύγματα της αποστολής αυτής, για την πρόοδο που είχε σημειωθεί. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη έλαβαν μία απόφαση πριν από λίγο καιρό να κλείσουν ε, την αποστολή αυτή μέχρι το τέλος του έτους. Επί του παρόντος προσπαθούμε να δούμε τι συνέχεια θα μπορούσε να δοθεί σε αυτή την αστυνομική αποστολή. Έρχεται λοιπόν την κατάλληλη στιγμή η δική σα συζήτηση, καθότι ε, η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει την Παρασκευή προκειμένου να δοθεί περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τον μηχανισμό που θα αποτελέσει μία συνέχεια τελικά για την αστυνομική αυτή αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Για να ταινίσουμε όμως το μέλλον θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το παρόν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τα επιτεύγματα της αποστολής αυτής, τι πρόοδος έχει σημειωθεί στο Αφγανιστάν. Ξέρετε ότι εκτελούμε μία εντολή που έχει να κάνει με συγκεκριμένε πτυχές μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει να κάνει επίσης με την επαγγελματοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων του Αφγανιστάν και συνεργαζόμαστε και με άλλους σημαντικούς παράγοντες που προσπαθούν και αυτοί στα πλαίσια των εντολών τους να συμβάλλουν. Μετά από 9 χρόνια λοιπόν η πρόοδο που είχε σημειωθεί από τι αφγανικέ αρχέ στα πλαίσια τη εντολή αυτή είναι πραγματική, είναι ρεαλιστική, αλλά πολλέ φορέ τα αποτελέσματα είναι μεικτά και εύθραυστα. Θα ήθελα καταρχά να αναφερθώ στην πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν. Έχει γίνει μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση. Έχουμε δει ότι όντω υπάρχουν νέε ικανότητε σε στρατηγικό επίπεδο και έχει αναπτύξει το Υπουργείο αυτό περισσότερε ικανότητε διοίκηση τη αφγανική αστυνομία τα ακόλουθα σημεία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μη στρατιωτική αστυνόμευση στο Αφγανιστάν. Έχουν προσταθεί περίπου 130 νέα όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών για την μη στρατιωτική αστυνόμευση και το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιε μονάδε σε όλε τι επαρχίε τη χώρα. Επίση, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε συγκεκριμένε πολιτικέ, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ για οποιαδήποτε βιώσιμη προσπάθεια γίνεται όσον αφορά για παράδειγμα μια πολιτική που έχει να κάνει με την ε, κοινοτική αστυνόμευση, με το θεσμό τη ε, ε, τοπικής αστυνομίας και στα πλαίσια της πολιτικής αυτής έχουμε και την υποστήριξη μονάδων οι οποίες αρχίζουν και να αναπτύσσονται όλο και περισσότερο σε επαρχίες της χώρας. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα πρότυπα λειτουργίας για την αστυνομία. Έχει υπογραφεί μια σχετική συμφωνία. Υπάρχει πλέον περισσότερο συντονισμό μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα και των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να γίνεται διερεύνηση ποινικών υποθέσεων, όπω συμβαίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Απαιτείται λοιπόν μια τέτοια συνεργασία μεταξύ Γενική Εισαγγελία και αστυνομικών δυνάμεων. Φέτο είδαμε ότι εγκρίθηκε και ένα μνημόνιο για τον Ombudsman, το διαμεσολευητή όσον αφορά την αστυνομία και τη λειτουργία τη αστυνομία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι περιπτώσει εκείνε που μπορεί να έχουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τι αστυνομικέ δυνάμει και έχουμε και μεταρρυθμίσει όσον αφορά την αστυνομική ακαδημία και τα προγράμματα κατάρτιση προβλέπονται από αυτήν. Όσον αφορά τις, ε, τα πρότυπα, τα ε, επιχειρησιακής διαδικασίας για την αστυνομία έχουν εγκριθεί κάποια νέα πρότυπα στα πλαίσια της αποστολής αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στα πρότυπα αυτά επιχειρησιακής λειτουργίας της αστυνομίας, τα οποία ισχύουν σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και στο Αφγανιστάν. Η λοιπόν θεωρείται πλέον ένας εταίρος αξιόπιστος από την αφγανική πλευρά η αποστολή αυτή έχει ε, προσελκύσει όλο και περισσότερη συμμετοχή από την αυγανική πλευρά τελευταία χρόνια και όπως ε, είπατε και εσείς και όπως είπε και ο διοικητής αποστολής αυτής τον Ιούνιο, καταφέραμε τα επιτεύγματα αυτά σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και αντίξω περιβάλλον. Βέβαια, οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν μπορούν να αποκρύψουν τις προκλήσεις που εκκρεμούν ακόμα για τις αφγανικές αρχές και για τη διεθνή κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό να μεταρρυθμιστεί το Υπουργείο Εσωτερικό, να γίνει μια επαγγελματοποίηση πλέον των αστυνομικών δυνάμεων του Αφγανιστάν. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί όλο ο τομέα ασφάλειας σε μια χώρα η οποία βρίσκεται ακόμα σε καθεστώς πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια κενά, δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη πρόοδος όσον αφορά την λειτουργία της αστυνομίας επιτόπου δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των πολιτών η νέα αυτή αφγανική αστυνομία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον κράτους δικαίου. Υπάρχουν ακόμα υψηλά επίπεδα διαφθοράς στη χώρα και σίγουρα το περιβάλλον ασφαλείας στο Αφγανιστάν είναι ακόμα ιδιαίτερα δυσχερές, καθότι η χώρα επισήμως βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση πολέμου και οι αστυνομικέ δυνάμεις προσπαθούν όλο και περισσότερο να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη χώρα. Όλα αυτά επηρεάζουν σαφώ κάθε προσπάθεια που γίνεται για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στι ίδιε αστυνομικέ δυνάμει. Πώ έχουν τώρα τα πράγματα. Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί η αποστολή αυτή. Αυτό έχουν αποφασίσει τα κράτη-μέλη. Η πρώτη φάση ήταν να κλείσει αυτή η γραμμή επιχειρησιακή που είχε να κάνει με το κράτος δικαίου. Αυτό συνέβη ήδη στα τέλη του 2015. Αυτή τη στιγμή ο ειδικό απεσταλμένο Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει συνέχεια στι δραστηριότητε αυτέ. Προβλέπεται όμω και μια σταδιακή αποχώρηση και σε κάποιου άλλου τομεί αποστολή. Υπάρχει ήδη μία ε, συγκεκριμένη ομάδα η οποία ασχολείται με, την, ε, το κλείσιμο και με την ε, διάθεση, αν θέλετε, των περιουσιακών στοιχείων των, της αποστολής αυτής. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Ξέρετε ότι η διάσκεψη των Βρυξελών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Αφγανιστάν με 5,2 δισεκατομμύρια τα οποία προβλέπονται ως χρηματοδότηση τα επόμενα τέσσερα χρόνια και όντως καταφέραμε να φτάσουμε σε 15,2 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2017-2020. Αναφέρομαι δηλαδή στις δωρές οι οποίες γίνανε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής των Βρυξελών. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο της μη, μη στρατιωτικής αστυνόμευσης. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη στους εμπειρογνώμονες της Καμπούλα και θέλουμε να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και την αστυνομία του Αφγανιστάν που θα είναι οι βασικοί μα συνομιλητέ. Η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιμείνει σε κάποιου τομεί όπου θεωρούμε ότι χρειάζονται οι Αφγανοί περισσότερο τη δική μα υποστήριξη και παροχή συμβουλών. Αυτό κάνουν και οι υπόλοιποι διεθνεί φορεί που βρίσκονται στο Αφγανιστάν και έχουμε ήδη καταλήξει στους τομείς συνεργασίας με την αυγανική πλευρά. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προδικάσουμε την απόφαση των κρατών μελών που θα συζητήσουν το ζήτημα αυτό στο τέλος της εβδομάδας όπως σας είπα. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την αυγανική πλευρά σε τρεις τομείς. Πρώτον, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ηγετική θέσης και λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ΟΜΑΙ, μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και καλύτερη, και καλύτερη επαγγελματικοποίηση της Αφγανικής αστυνομίας με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που θα έχουν να κάνουν με την τοπική αστυνόμευση και με καλύτερη συνεργασία μεταξύ εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων για τις εγκληματολογικές έρευνες και θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε να διαρευνούμε περισσότερο περιπτώσεις διαφθοράς και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και να προωθήσουμε το ζήτημα της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στις αφγανικές αστυνομικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, η αυγανική πλευρά θα συνεχίσει να εξαρτάται από την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα συνεχίσει το έργο το οποίο έχει, είχε ήδη ξεκινήσει η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Θέλουμε απλώς να δούμε ποιον ακριβώς μηχανισμό θα εγκρίνουμε για την μικρή αυτή ομάδα των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που θα παραμείνει στο Αφγανιστάν. Ολοκληρώνω σε σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέρκα. Um, Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, κυρία Πρόεδρε, για τη σημερινή σας ε, συνεδρίαση. Πρώτα-πρώτα, Είπαμε για το ότι θα πρέπει να θυσιαστεί η Γιούπολ. Το προσωπικό, η προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι υπέστησαν πάρα πολλέ απώλειες ε, για απώλεια ανθρωπίνων ζώων κατά την αποστολή τους και όλοι όσοι εκεί αποσπάστηκαν και απασχολήθηκαν εκεί ήταν Ευρωπαίοι ή Αφγανοί. Και όλοι αυτοί ε, ασχολήθηκαν με μεγάλη φιλοτιμία με τη δουλειά τους και θα πρέπει όλους αυτούς να τους τιμήσουμε για τη διαδρομή τους όλα αυτά τα χρόνια. Και θυμάμαι όλους εκείνους τους πολίτες, ε, τους Αφγανούς, οι οποίοι ε, σκοτώθηκαν από κάποια επίθεση που ήταν κατά τη Γιούμπολα, αλλά τελικά την πλήρωσαν εκείνοι. Το 2010 ασχολήθηκα σαν αναλυστής και κατόπιν ε, ήμουν το νούμερο 2 σε κάποια φορέα συντονισμού για την UPOL ε, και την ε, αστυνομική της ε, αποστολή. Επίσης είχαμε συμμετάσχει σε αποστολέ του ΝΑΤΟ, κάποια ομάδα που πρόκειται να του γίνει η Γερμανία και να ξεκινήσουμε να δούμε το ευρύτερο τοπίο, να δούμε σήμερα πώς έχει η κατάσταση. Όσον αφορά το μέλλον της χώρας, ακόμα υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα. Το 2015 ήταν μια χρονιά όπου χάθηκε και άλλο έδαφος και από το 2001 έτσι έχουν πάει τα πράγματα για την κυβέρνηση και τους ε, συμμάχους. Και επίσης στο νότο κατέρευσε το μέτωπο και οι απώλειες ακόμα είναι ενισχυτικά μεγάλες. Στην άλλη μεριά υπάρχει είναι δύσκολη κατάσταση οικονομική στη χώρα, ε, συνεχίζεται η επιστάτευση. 23% ήταν οι απώλειες. Α, και μιλούμε για τραυματίες αλλά και λιποτάκτες. Όταν μιλούμε για τους εταίρους μας, στο Αφγανιστάν, την κυβέρνηση δηλαδή, μιλούμε για σχέσεις σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Αλλά βέβαια είναι πολύ ευάλωτη αυτή η εταίρη μας. και ο πρόεδρο τη χώρα και ο πρόεδρο τη αντιπολίτευση και ο αρχηγό αντιπολίτευση τέλο πάντων βρίσκονται σε συνεννόηση με κάποιο συμβασμό. Οπότε έτσι ε, γίνεται η διακυβέρνηση της χώρας με, τα, με κάποιο φορολογικό σύστημα που μάλλον είναι διεφθαρμένο ε, ασκείται η φορολογική πολιτική και επίσης το ίδιο συμβαίνει διαφορά δηλαδή και στις ε, ενοπλές δυνάμεις. Ακόμα δηλαδή δεν υπάρχει αξιοκρατία όσον αφορά την αστυνομία και τις ενόπλες δυνάμεις. Βεβαίως όμως υπάρχουν και οι αξιόλογοι αξιωματικοί και στα δύο σώματα. Δεν λείπουν τα κίνητρα για αυτούς τους αξιωματικούς. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις επίσης για όλες τις πρωτοβουλίες και έχουμε συνεχείς άνασχηματισμό στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το καλοκαίρι ορίστηκε καινούριο ε, Υπουργό Εξωτερικών και από το 2001 είχαμε τη Βόρεια Συμμαχία οπότε και στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν κάποιοι πάρα πολύ αξιόλογοι. Δέκα με έντεκα ήταν πολύ καλός ε, υπουργό ο κ. Μοχάμετ. και ταξίδευσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι ο σύμβουλος του ΝΑΤΟ σημείωνε στο χάρτη που πήγε ο υπουργό και πήγε παντού στο βορρά, δεν είναι ασφαλής περιοχή. Τέλος πάντων δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συνέπεια στη δράση της κυβέρνησης. Προσπαθούν να, να υπάρξει εμπιστοσύνη από πλευράς της χώρας. Αλλά είπαμε ότι υπάρχει αυτού του είδους η διεφθαρμένη φορολόγηση και επίσης στην κυβέρνηση υπάρχουν πολλές φράξεις, πολλές ομάδες. Και Ακόμα και στα πλαίσια και στους κόλπους του ίδιου Υπουργείου υπάρχουν πολλές ομάδες που δρούν αυτόνομα. Τώρα από πλευράς υποστήριξης από τον ΝΑΤΟ. Στη χώρα ξεκίνησε η αποστολή σαν αντιτρομοκρατική, συμβουλευτική, επικουρική της ε, ε, μη στρατιωτικής αποστολής. Και όμως υπήρξε και βοήθεια από αέρος και αυτό βοήθησε στο να μην προχωρήσουν ακόμα περισσότερο οι Ταλιμπάν. Όμως είπαμε ποια είναι η αντισχετική τάση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο ισχυρή η αφγανική αεροπορία. Οπότε τα, τα πράγματα γίνανε δύσκολα για την κυβέρνηση, ζητούσαν από εμάς ε, αεροπορικές επιδρομές και το θέμα ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα. Θα πρέπει η αφγανική αεροπορία να αναβαθμιστεί και να τα καταφέρει. Ο πλευρά τώρα Αμερικανική πολιτική φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγον η και η στρατηγική των ΕΠΑ μπορεί να χωριστεί σε τρει άξονε. Πρώτα-πρώτα η, δύναμη για να αντικαταστήσει τι δύναμη του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, του να υπάρχουν κάποιε ε, ε, ε που να δουν τοπικά και τρίτον η ε, συνδιαλλαγή με τους ε, Ταλιμπάν. Και στους τρεις άξονες αυτούς και στα τρία μέτωπα αυτά απέτυχε η Αμερικανική πολιτική. και σε επίπεδο επιμελητίας, ε, προμηθειών, διοίκησης και προγραμματισμού. Όλα αυτά είναι προβληματικοί τομείς, όπως διαπιστώνεται. Και όσον αφορά την την αυγανική αστυνομία πολλές φορές αντί για σεβασμό, την χάνει φόβο σε πολλά μέρη στη χώρα και πολλές φορές ε, η αστυνομία παίρνει το πλευρό κάποιων συγκεκριμένων φατριών ή οικογενειών οπότε όποιος είναι έξω από ένα συγκεκριμένο κύκλο από συγκεκριμένη φατρία ε, έχει πρόβλημα. Οπότε υπάρχει θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά δεν ε, βρουν ε, σαν διοικητική αρχή, σαν αστυνομία, είναι κάτι σαν φύλακες, ε, στατικά συμπεριφέρονται και, ε, όπω είπαμε, επικουρούν τους τοπικούς πολέμαρχους. είπα είχε εξοδέψει πάνω από 60 δις δολάρια για τις ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πολλά χρήματα. Και όπως είπαμε, για αποδιοίκηση, προγραμματισμό κλπ. Εκεί δεν προχώρησε η υπόθεση. Και αυτό διότι υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση ε, όσον αφορά τους πολιτικούς και την πολιτική στην χώρα. Ο καθένας περασπίζεται το δικό του μετερίζει. Ο κάθε πολιτικός παράγοντας. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε εδώ εθνικές ανάγκες. Εκεί η κάθε ομάδα φροντίζει τα δικά της συμφέροντα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντική η στην αστυνομικών και στρατιωτικών Αφγανών. Έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες απώλειες και παρά όλα αυτά τα προβλήματα επιμελητίας ε, έχουν καταφέρει πολλά. Έχουν κρατήσει τις θέσεις τους σε πολλά σημεία. Ούτε καν αρκετά νοσοκομεία δεν υπάρχουν για τους τραυματίες. Πάρα πολλές φορές οι ευγενικές μονάδες έχουν περικυκλωθεί και έχουν αποδεκαριστεί και πολλές φορές εμείς βάλουμε πολύ ψηλά τον τύχη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ζητούμε από τους Αφγανούς αυτά τα οποία ζητούμε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που είναι πολύ πιο καλοζωισμένοι εκεί οι στρατιώτες. Άρα βλέπουμε ότι κλιμακώνεται εκεί η αντιπαράθεση και δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα πάνε προς σωστή κατεύθυνση γιατί Γιούπολ τώρα. Τρία σημεία. Πρώτο πρώτο, Το προσωπικό για την ιεραρχία. Δεύτερον. Στόχοι. Και τρίτον. Το Υπουργείο των Εσωτερικών και Αστυνομία. Επίσης, το κατά πόσον ε, συμβάλλει σε κράτος δικαίου η υπηρεσία αυτή. Από την αρχή υπήρχαν προβλήματα αλλά το ότι συνέχεια άλλαζε η εντολή αυτό δεν βοήθησε. Σήμερα να Βρυξέλλες αντί για το ίδιο το Αφγανιστάν. Συνέχεια με προσαρμογή της εντολής τους. Και το 2009 υπήρχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα βοηθούσε και τον ΝΑΤΟ. Ε, ουσιαστικά όμως πολλές φορές γινόταν απλώς κατανομή του οικονομικού βάρους. Μπορεί να είχαμε στη μία πόλη καναδική αποστολή ε, και αλλού να είχαμε βρετανική. Πολλές φορές όμως ε, υπήρχε προτίμηση της προτεραιότητες του ΝΑΤΟ που ήταν το πλαίσιο στο οποίο κινούνται παρά προσήλωση στις προτεραιότητες της γιου πολιτιστικής. Οπότε συνέχεια υπήρχε μεταστροφή στο τι στόχοι επιδιώκονται. Άρα τα χρήματα που πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιάσαν τόπο. Ακόμα και στο στρατηγείο υπήρχαν ε, κάποιοι αστυνομικοί Ευρωπαίοι και πιεζόντουσαν να κάνουν διάφορα πράγματα ε, αντιτρομοκρατικής φύσης πολλές φορές. Οπότε βέβαια και εξοδεύαν πολύ χρόνο γι' αυτό. Και χρησιμοποιούσαν τη Γιούπολη για αυτές τις άλλες δραστηριότητες κάποιες φορές. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Και το ΝΑΤΟ δεν το αντιμετώπισε αρκετά. Οι χώρες δηλαδή που συμμετέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποστολή δεν προσπαθούσε να τα διορθώσει, αλλά μια που ε, κυρίαρχο φορέα ήταν το ΝΑΤΟ, είχε πρόβλημα η Γιούπολ για να τα καταφέρει. Πολλέ φορέ. Το θέμα τη εντολή τώρα. Προσπάθησε η Γιούπολ να ασκήσει έργο μη στρατιωτική αστυνομία, να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ και με τι αφγανικέ αρχέ. Και θυμάμαι με το κοινό επιτελείο υπήρχε ο στρατηγός Ροντρίγκε και μίλησε για το πόσα απόλυση έχει η οργανική αστυνομία και κάποιος από τη Γιουπολή δεν μας νοιάζουν τώρα οι δολοφόνοι, μας νοιάζουν οι αστυνομικοί. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί είχαν πάρα πολλές απόλυες αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά και τους άγγιγε το θέμα της αεροπορική υποστήριξης. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ανέστητοι. Ας θυμηθούμε και τον Τρότσκι, όπου έλεγε ότι μας νοιάζει η αστάθεια στη χώρα η εξέγερση, αλλά ασχολείται η αστάθεια με μας. Οπότε θα πρέπει κανείς να προσαρμόζεται, να προσπαθεί να καταλάβει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ε, αστυνομία της χώρας στα επικίνδυνα σημεία που δρούσε. Άρα δεν ήταν πάντα ζήτημα προτεραιότητας τούτο. Καμία σχέση με το τι γίνεται στο Βασίλειο και στη Σουηδία, ας πούμε, το πρώτο θέμα ήταν κανείς να μείνει ζωντανός για να μπορέσει να υπηρετήσει και την επόμενη εβδομάδα. Άρα τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλαμε. Κατανοητό αυτό. Άρα δεν ήμασταν ίσως τόσο λογικοί. Και θα έπρεπε για να αξίζει η παρουσία μας εκεί να μπορέσουμε να τους στρέψουμε την προσοχή τους εκεί που έπρεπε στο σημείο σημείο της χώρας επίσης ο στρατηγικός ρόλος η επιρροή μας στο Υπουργείο Εσωτερικών Πολλέ φορές υπήρχαν σύμβουλοι, υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι είχαν επαφή με τον Υπουργό γιατί το ΝΑΤΟ τελικά και είπα χρηματοδοτούσαν. Εκείνοι συνόδευαν τον Υπουργό μετακίνηση του. όχι εμείς. Άρα, αντί να ασχολούνται με τα θέματα αστυνόμευση που ενδιαφέραν εμά, ασχολούνται με το πώ θα πλαισιώσουν ή θα προστατεύσουν τον Υπουργό Συμμετοκίνηση. Άρα, πολύ εντατική δράση, αλλά δεν υπήρχε αποτίμηση του τι καταφέρνουμε τελικά με όλη αυτή την δραστηριότητα σε κάθε περιφέρεια. Η ISAF, το κοινό επιτελείο, ήταν ε, ε, βασική, βασικός φορέας, βασική υπηρεσία με το οποίο είχαμε επαφή. Μόνο αυτοί λοιπόν ασχολιόντουσαν με αυτό το move, shoot, communicate της, των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της Αφγανικής ε, Αστυνομίας. Οπότε είχαμε συλλήψεις και προμπή στην δικαιοσύνη από την αστυνομία. Όμως αυτή η κατάσταση δεν κράτησε πολύ δυστυχώς. Άρα η ISAF χρησιμοποιούσε την αστυνομία σαν ελαφρό πεζικό. Όμως, είπαμε αυτό δεν κράτησε πολύ. Και από πλευράς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, το οποίο επίσης ήταν αρμοδιότητα της Γιούπολ. Εντάξει, όσο ο εκπαιδευτής μένει εκπαιδευτής. Όμως, δυστυχώς αυτοί που εκπαιδεύαμε δεν παρέμειναν εκπαιδευτές. Και αυτό ήταν δύσκολο θέμα να το επιλύσουμε με τους εκεί εταίρους μας. σε ανώτατο επίπεδο και με ειλικρίνεια έπρεπε να λύθει το θέμα. Και σωστή λύση το να εξαρτήσει κανείς τη βοήθειά του από το να τηρήσει ο άλλος τα συμπεφωνημένα. Οπότε είχαμε αστυνομικούς σε θέσεις συμβούλων. Οι μέντορες του Υπουργείου που είναι μια έννοια και μια λέξη απέσια και προσβλητική, αλλά τέλος πάντων είχαμε τους στρατηγούς που καμιά φορά πέραν συμβουλές από απλούς αστυνομικού. που ποτέ δεν είχαν κάνει αυτή τη δουλειά, οι οποίοι στη δουλειά τους αυτοί οι αστυνομικοί ήταν καλοί. Ποτέ όμως δεν είχαν πάει στο εξωτερικό και κάποιοι από αυτούς δεν είχαν ξαναπαντήσει το πόδι τους σε Υπουργείο. Πάντως, τέλος πάντων, στην ε, Ευρώπη κάθε αστυνομία έχει διαφορετικά πρότυπα, διαφορετική οργάνωση. Οπότε και για την υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, αυτό είναι πρόβλημα για τις αποστολές. Τι θα κάνει μόνος θα κάνει ό,τι έκανε στη χώρα του. Οπότε, πώς θα δράσει η αποστολή όταν πολλοί αστυνομικοί από διάφορε χώρε είναι στην ίδια αποστολή. Μέχρι τώρα σας είπα τα σκούρα. Για να δούμε όμως υπάρχουν και αισιόδοξα και αξιόλογα σημεία και επιτεύγματα. Πρώτα-πρώτα συγκεκριμενοποιήθηκε η εντολή της Γιούπολης επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένα σημεία, φύγαμε από τα ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ, ε, ασχοληθήκαμε με την Αστυνομική Ακαδημία και τελικά κάτι καταφέραμε και αφήσαμε σαν κληροδότημα για την αυγανική αστυνομία για το μέλλον. Άρα, τα εύσημα πάνε σε χώρες μέλη για το τι έκαναν. Είχαμε 70.000 ε, Αφγανούς αστυνομικούς οι οποίοι ποτέ δεν ε, έκαναν αστυνομία όπως την ξέρουμε ήταν απλώς ε, κάτι σαν σεκιουριτάδες. Επίσης ασχολήθηκαν και με ποινικέ υποθέσεις, εγκλήματα δηλαδή. Οπότε, αν βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα, τότε νομίζω ότι η αυγανική αστυνομία μπορεί να ωφεληθεί από όσα κάναμε εκεί. Πάντως, δυστυχώς, για πολιτικούς λόγους, από πλευράς διοικητικής είναι αδύναμο το Υπουργείο Εσωτερικών, παρά το ότι υπάρχουν εκεί ικανοί υπάλληλοι. Αλλά συνέχεια καπελώνονται, αγνοούνται σε αυτό το οποίο λένε για μικροκομματικούς πολιτικούς λόγους. Ευτό και δεν έχει δημιουργηθεί και ένα σώμα επαγγελματικών, ας πούμε, ε, αξιωματικών και υπαλλήλων. Είχαμε επομένω εμείς ως προτεραιότητα την καταπολέμηση τη διαφθορά. Όταν όμως απειλείται η ζωή του επικεφαλής του Υπουργείου για κατά διαφθοράς από τον Υπουργό, δεν λέγαμε τίποτα. Οπότε και αυτός δεν ενδιαφέρονταν να κάνει τη δουλειά του, αφού του απειλούσαν την ζωή, επειδή τα πήγε καλά στις έρευνες. Οπότε στην εκπαίδευση λέγαμε ασχοληθείτε με την καταπολέμηση της διαφθοράς, συνέχεια ε, επειδή υπήρχε καπέλωμα των υπηρεσιών και κλείσιμο, κάναμε καινούργιε υπηρεσίε και λέγαμε ότι τώρα ήρθε η ώρα κάτι να γίνει, θα πρέπει να προβάλλουμε κάποιο ζήτημα και στους Αφγανούς εταίρους και στο ΝΑΤΟ, οπότε η Αμερικανική Πρεσβεία το βλέπει αυτό και ήταν δύσκολη η σχέση τους με την ε, εκπαιδευτική αποστολή και ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές ε, είχαν στο μυαλό τους το ήταν εκεί για πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Είμαι εδώ για έξι μήνες, αλλά θα πρέπει έτσι να ενεργήσω. Δεν, δεν λάβαναν υπόψη το καλό της ε, αποστολής. Αν δεν μπορούν να πιάσουν τόπο τα λεφτά που δίνει κανείς, καλύτερα να μην τα δίνει. Οπότε αυτή η σύντομη θητεία του προσωπικού δεν ωφελούσε. Θεωρούσαν και τους εξόριζαν και τους στέλνουν στην πατρίδα και για τις Βρυξέλλες αυτό και λέγαμε ότι μήπως πρέπει να μπει ο ιδιωτικό τομέας και εγώ πολλές φορές είχα αμυντική στάση στην αποστολή προσπαθώντα να κάνω το καλύτερο ακριβώς γιατί υπήρχαν εμπόδια πολιτικής φύση πέρα από τον έλεγχό μου. Επομένως και στο Υπουργείο Εσωτερικών και αλλού είχαμε αυτά τα πολιτικά προβλήματα, προσπαθούσαμε να τα κανονίσουμε. Ε, δηλαδή προηγείται το, το, πολιτικό θέμα και μετά το τεχνοκρατικό. Άρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ας πούμε διαμεσολαβητή, αλλά είχαμε όλες αυτές τις ε, απειλές. Άρα πώς κανείς να δουλέψει αν δεν συμβαίνει τίποτα. Άλλο πρόβλημα. Υπήρχε άγνοια του Ισλαμικού δικαίου στο Αφγανιστάν. Παρά το ότι είναι αυτός ο, ο νόμος που ισχύει. Παρά λοιπόν το ότι πάρα πολλοί από το προσωπικό ε, είχαν δράσει σε όλο τον κόσμο, δεν καταλάβαινε τα το του Ισλαμικού δικαίου. Αυτό δηλαδή που είναι δεδομένο για τους Αφγανούς. Προσπαθούσαν λοιπόν να θεσπίσουν διαφορετικό δίκαιο, οπότε υπήρχε κάποιο είδους ασυνέπεια συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και για το, δικαστήριο, για τη δικαιοσύνη. Δεν ξέραμε πώς να συνεχθούμε, να έχουμε μια κοινή γλώσσα με τους αστυνομικούς. Οι περισσότεροι των οποίων ακόμα και οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν ξέρανε τι πάει να πει η ποινική δικονομία, δεν ξέρανε πώς να δουλέψουν επί τη βάση κάποιου ποινικού κώδικα. Είχαν δηλαδή δυνατότητες, αλλά δεν έπιαναν τόπο. Και στέλναν κόσμο στο δικαστήριο, στη δικαιοσύνη. Όμως και στην εισαγγελία υπήρχε θέμα διαφθοράς. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε, αλλά ήταν τόσο βαθιά και ε, ευρία η διαφθορά. Και ακριβώς και με την άγνοια του Ισλαμικού δικαίου δεν μπορούσαμε να δράσουν καλά. Η Γιούπολ σε μια χώρα στο Αφγανιστάν είχε έργο πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολλοί προσπάθησαν πάρα πολύ για να βελτιωθούν τα πράγματα. Γι' αυτό και η Γιούπολ θα πρέπει να αξίζει συγχαρητηρίων. Και δεν μιλάμε τώρα για στρατιωτικούς. Μιλούμε για κάποιους ε, οι οποίοι αποσπάστηκαν εκεί για πρώτη φορά στην σταδιοδρομία τους. Και τα πήγαν πάρα πολύ καλά. πολλές εγκληματικότητας και εκεί καλές επιδόσεις. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν και την παρούσα και τη μέλουσα αφγανική κυβέρνηση. Όμως θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κάποια διοίκηση, κάποια αστυνομία με επαγγελματικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλοί εργατικοί και ικανοί Αυγανοί, αλλά όλα αυτά είναι πολύ βραχυπρόθεσμα για, για τους λόγους που είπαμε. Και όσον αφορά αυτό το civilian planning το ίδιο, θα πρέπει να δούμε το κατά πόσον κανείς με λιγμούς θα μπορέσει να ξεπεράσει τα πολιτικά προβλήματα από πλευράς τεχνοκρατικής ή αν θα κάνει κάποιες άλλες αλλαγές που θα κρατήσουν περισσότερο. Υπάρχει πρόβλημα στο Υπουργείο και άρα δεν ξέρω θα ανησυχώ για το μέλλον της Αφγανικής Αστυνομίας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πολιτική ζήτηση που θα πρέπει να γίνει και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τάξουμε κάποιες προτεραιότητες και αν θέλουμε να χρηματοδοτούμε θα πρέπει να απαιτούμε σοβαρές βελτιώσεις. Διαφάνεια στον προϋπολογισμό, στην διαχείρισή του, να ζητήσουμε να μας αναφέρουν σχετικά με το πώς απορροφούνται τα κονδύλια και θα πρέπει οι εκπαιδευτές να μένουν εκπαιδευτές, αυτοί που εμείς εκπαιδεύουμε και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η Ιούπουλ θα έχει βοηθήσει για να υπάρχει μια νέα γενιά θεσμών στη χώρα και που να διακρίνεται από επαγγελματικότητα. Δεν το αποκλείω. Οπότε ε, επιμένω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το civilian planning capability και η UPOL ε, ε, πήγαν πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις εισαγωγικές παρουσιάσεις και τώρα θα αρχίσει η συζήτηση και θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον επικεφαλής της αποστολής για το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρό... κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν που οργανώσατε αυτό, αυτή την ε, συνάντηση, την ακρόαση και καλέσατε ειδικού εμπειρογνώμονες που ακούσαμε μεγάλη μας χαρά. Ε, πρόκειται για ένα σημαντικό συμβάν γιατί είχαμε μια ιδιαίτερος ε, πετυχμένη συνάντηση κορυφή του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύνοδο κορυφή όσον αφορά τι αποφάσεις για το Αφγανιστάν, καθώς και τον Οκτώβριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει λοιπόν το θέμα της συνέχισης και των ενδεχόμενων αλλαγών ε, σε σχέση με το Αφγανιστάν και τη δική μας αποστολή γιατί ε, πραγματικά να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ε, χρηματοδότηση και τα δις τα οποία υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη ε, στο Αφγανιστάν τα οποία ε, μας υποχρεώνουν να προβληματιστούμε και να δούμε ε, ποιοι θα είναι οι νέοι στόχοι λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω ε, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της ε, προηγούμενης εμπειρία μας. Ε, ένα πράγμα είναι σαφές. Δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε το Αφγανιστάν στη μοίρα του και η δική μας δέσμευση είναι απολύτως θεμητή και έχει μια στέρεη ηθική βάση. και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη συνέχισή τη. Αλλά ακούγοντα του απειρογνώμονε έχω πράγματι ορισμένε επιπρόσθετε ερωτήσεις για αυτού, αλλά και για όλου μας. Επικεντρώθηκαν αρκετά στην εκτελεστική εξουσία στο Αφγανιστάν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός, κοινοβουλευτική εξουσία σε αυτή τη χώρα. Όχι συχνά, αλλά από καιρού καιρών υπάρχουν κάποιες ε, επισκέψει γίνονται στο Αφγανιστάν. Το ερώτημά μου έχει στο εξή. Τι γίνεται με, την, με το Αφγανικό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις ε, πρόοδους των μεταρρυθμίσεων στις οποίες αναφερθήκατε. Έχετε κάποια στοιχεία σχετικά και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς τους πολιτικούς. Ε, παρόλο που η διάκριση των εξουσιών στο Αφγανιστάν είναι διαφορετική από ό,τι εδώ. Και ορισμένες φορές το Κοινοβούλιο δεν έχει ε, ε ισχύ λήψης αποφάσεων. Ε, ωστόσο, σε ποιο βαθμό την προσεχή περίοδο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την ισχύ του Κοινοβουλίου, την κοινοβουλευτική εξουσία ε, και επίσης τις κοινοβουλευτικές ε, εξουσίες αρμοδιότητες ελέγχου, άσκηση ελέγχου, προκειμένου να αποφύγουμε τους κινδύνους ε, διαφθοράς και της αναπολετελεσματικής χρήσης των κονδυλίων των διεθνών δωρητών για το Αφγανιστάν. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει εξής. Ε, δεν έχουμε μια αποτελεσματική δίκηση στο Αφγανιστάν και δεν μπορούμε να αναμένουμε κάποιες ε, ε, εξελίξεις, προόδους μάλλον σε διάφορους τομείς. Θεωρείτε ότι το μοντέλο της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία συνεχώς βελτιώνεται, ε, μπορεί να ισχύσει με περισσότερα κονδύλια ή ε, θα έπρεπε να υπάρξει ένα διαφορετικό μοντέλο, όπως είπατε. Δηλαδή, ενδεχομένως θα έπρεπε να εντάξουμε τους δικούς μας εμπειρογνώμονες περισσότερο στις ε, ομάδες των Αφγανών με ένα διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε όχι να τους συμπληρώνουμε απλώς, να κομίζουμε τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη, αλλά για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια να ενταχθούμε και εμείς ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε μεταβολές στην ουσία των πραγμάτων τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένω να οδηγήσουν σε μια καλύτερη διακυβέρνηση γενικά. Τέλος, όσον αφορά τα ελλείμματα στους ε, θεσμούς, την αδυναμία μάλλον των θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι φιάλτη στον, στο Αφγανιστάν. Πολύ συχνά έχουμε συχνές ε, αλλαγές των διαφόρων κλιμακίων της εξουσίας και ε, δεν μας επιτρέπουν περιθώριο αισιοδοξία σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία εφόσον εφαρμοστούν ε, αναμένουμε να βελτιώσουν το σύστημα αυτό καθ' αυτό. Πώς αξιολογείτε την γενική, ε, το γενικό επίπεδο, την κατάσταση των ε, θεσμικών οργάνων που διακυβερνούν τη χώρα. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιους δείκτες που θα μας οδηγούσαν σε κάποια συμπεράσματα σχέση με το δικό μας πρόγραμμα συνδρομής και δική μας προσέγγιση στη χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να αναλύσετε εδώ την κατάσταση και να μας παρουσιάσετε αυτά τα συμπεράσματα. Ελπίζω ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να αντιλήσουν από τη σύντηση αυτή και από τη δική σας εμπεριγνωμοσύνη στοιχεία τα οποία ενδεχομένω θα μπορούσαν να επιφέρουν βελτιώσεις όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, αλλά και στο ίδιο το Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκάλαρ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πάρτε τα, τα ακουστικά σας, γιατί θα μιλήσω γερμανικά. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ τους δύο ε, ε, ε εμπειρογνώμονες ήταν πραγματικά κάποιες ρεαλιστικές και τίμιες ε, παρουσιάσεις ε, που κατά κάποιο τρόπο μας αφήνουν αμήχανους. Ε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τους δικούς μας εμπειρογνώμονες και τους αστυνομικούς που μετέβησαν στη χώρα, γιατί πραγματικά τα κινήτρά τους ήταν ισχυρά. Ε, πήγαν την καλύτερη δυνατή θέληση, αλλά προσέκρουσαν σε κάποιες δομές, οι οποίες παρουσιάστηκαν εδώ, οι οποίες είναι κατετμημένες, υπάρχει μια πολυδιάσμαση, δεν είναι η γνωστή σε εμά διάρθρωση όπου υπάρχει ένα υπουργείο, υπουργό, η πολιτική γραμμή κλπ. Αλλά εκεί στο Αφγανιστάν υπάρχουν οι φύλαρχοι, οι πολέμαρχοι, υπάρχουν ε, οι πολιτοφυλακές και θα πρέπει να δει κανείς ποιος ανήκει πού, ποιος δηλώνει πίστη σε ποιον ε, φύλαρχο, σε ποια ομάδα, σε ποιο πολέμαρχο κλπ. Ε, και δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν όλα αυτά μπορούν ε, να έχουν νόημα, οι δικές μας προσπάθειες εννοώ. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα εν σχέση με το πώς θα πρέπει να διαμορφώσουμε τη μελλοντική μας στρατηγική. Αλλά να γνωρίσαμε πρώιμα ότι οι αρχικές μας προθέσεις ε, δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν γιατί είχαμε πέντε αλλαγές εντολών και αυτή πραγματικά ήταν μια αντίδραση στην, ε, στις τη της πρώτης, της μετέπειτα εντολής. Και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε κάθε φορά την κατάσταση. Αλλά έτσι όπως ε, πράγματι υπόθηκε, θα πρέπει να, είναι, να υπάρχει καταρχήν μια, ε, σαφήνεια σε πολιτικό επίπεδο, να είναι ξεκάθαρη η πολιτική στόχη, πολιτική, πριν εμείς μεταβούμε εκεί και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να πραγματοποιήσουμε κάτι. Ε, πιστεύω ότι ε, αυτό το οποίο επίση ε, μπορεί να θεωρηθεί ως δίδαγμα ή συμπέρασμα είναι το εξή ότι ως διεθνής κοινότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τις ΗΠΑ και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να έχουμε μεταξύ μας καλύτερο συντονισμό ε, και αν εκεί υπάρχει μια ισχυρή, μια αστυνομική αποστολή από τη ΣΥΠΑ, δεν μπορούμε εμείς να δρούμε εκ παραλίλου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος επιμερισμός των καθηκόντων, ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο ε, το που αποβλέπουμε και τι αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε. Εγώ συνολικά ε, γενικά μάλλον είμαι θλιμμένος από το αποτέλεσμα. Και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να καταλήψουμε τη ελπίδα εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση αυτοί οι οποίοι είναι επαρκώς ειδικευμένοι κάποια στιγμή να μπορέσουν να επιδράσουν θετικά στην πραγματικότητα της χώρας. Θα είχα ωστόσο και μία ερώτηση την εξής. Γιατί δεν πέτυχε τουλάχιστον εκεί επί τόπου να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της τοπικής αστυνομίας. Της αστυνομίας. Ε, community policing ε, αναφέρθηκε εδώ. Τι είναι αυτό. Είναι η τοπική αστυνομία ε, και γιατί δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει εκεί κάποια, κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η υπόθεση είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η διαίρεση σε διάφορες ε, φυλές, τότε η τοπική αστυνομία θα υπάγεται στον τοπικό φύλαρχο, στην τοπική φρατρία. Αλλά όταν άκουσα ότι μάλλον φοβούνται παρά σέβονται την τοπική αστυνομία, local police, αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουν αποσταλεί κάποιοι από την πρωτεύουσα, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ε, τοπικές συνθήκες, ε, ούτε προσωπικά, ούτε ανήκουν στην ίδια φυλή ενδεχομένως. Και αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση αν θέλει κανείς να έχει εμπιστοσύνη σε μια χώρα, τουλάχιστον ε, η τοπική αστυνομία να είναι από την ίδια περιοχή, να μιλάει την τοπική γλώσσα και να έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών της περιοχής. Αλλιώς ε, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Εγώ πραγματικά δεν έχω πλέον ψευδεστήσεις ε, μετά από όλα όσα άκουσα. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναγκόμες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ εδώ από την αρχή να ακούσω τις παρουσιάσεις, ωστόσο έχω τις εκθέσεις και το ερώτημά μου ε, ευθυγραμμίζεται με αυτά στα οποία αναφέρθηκαν ήδη οι συνάδελφοι. Ε, στη βάση της δικής μου εμπειρίας στο Αφγανιστάν το 2008 όταν ε, σχηματίστηκε η UPOL, ήταν στην αρχή της τα Σπάργανα και ακούσαμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τότε παραμένουν και σήμερα. Δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς μη επαγγελματική δομή αστυνομίας, απολύτως διεφθαρμένη, με μια απολύτως διεφθαρμένη δικαιοσύνη και πολύ αδύναμες ε, κυβερνητικές δομές. Ήταν λοιπόν ένα φιλόδοξο, πολύ μεγαλόπνο ε, πρόγραμμα. Τότε ήμουνα σε μια κυβερνητική αποστολή. Ίσως δεν ήταν αναγκαίος αυτός ο τύπος αστυνόμευσης στο Αφγανιστάν. Ενδεχομένως θα χρειαζόμαστε περισσότερο μια προσέγγιση τύπου χωροφυλακής. Όχι τη μη στρατιωτική αστυνομία, η οποία είναι γνωστή στις ευρωπαϊκές χώρες. Ε, ε, εσείς ε, συμπελάβατε όλα αυτά τα θέματα στην προσέγγισή σας. Ένα άλλο μείζον ε, πρόβλημα στο Αφγανιστάν ήταν ότι στις φυλακές του Αφγανιστάν ήταν ε, περισσότερες γυναίκες από εγκληματίες απλώς και μόνο επειδή είχαν ε, αποδράσει από τους συζύγους τους και απλούστατα αυτό που έκανε ήταν τους έβαζαν στη φυλακή. Έχει αλλάξει αυτό μετά από 8 χρόνια. Και ένα άλλο ερώτημα, οι πρόσφυγες. Εάν δει κανεί τα προσφυγικά στατόπεδα στην Ελλάδα ή στο Καλέ, ε, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πολλέ αφγανικές οικογένειες και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι Αφγανοί. Και πολλοί από αυτού, ε, εγώ είδα αγόρια 7 ή 8 χρονών. Πολλοί από τους Χαζάρα, από τη μειονότητα των Χαζάρα, η οποία ε, ε, υποφέρει τα πάνδυνα στο Αφγανιστάν την οποία ε, επίσης εκμεταλλεύονται σεξουαλικά οι ενήλικοι Αφγανοί, αυτούς τους ανηλίκους, τους χαζάρα ανηλίκους. Πολύ συχνά είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ε, κάνατε κάτι εδώ με την Αφγανική αστυνομία. Και μία τελική ερώτηση. Προβλέπετε να παίξετε κάποιο ρόλο στο όργανο το οποίο θέλει να συστήσει το Συμβούλιο. δίνοντας έμφαση στην πανιστοχή των ε, δύστιχων Αφγανών οι οποίοι έχουν αποδράσει και των οποίων η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου ασφαλής. Η κυρία Σαμπίνα Λόζινγκ, ε, παρακαλώ θα μιλήσω γερμανικά. Εγώ ε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετικά περιεκτική ανάλυση και την ε, φροντίδα που επέδειξαν εδώ οι συνάδελφοι τις ανησυχίες αυτές, τις δικές ανησυχίες συμμερίζονται όλοι εδώ στην αίθουσα. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα συμπεράσματα τα οποία θα έπρεπε να αντλήσουμε. Ο κύριος Γκάλαρ αναφέρθηκε στο φόβο που αισθάνονται οι κάτοικοι ε, από, ε, μπροστά στην αστυνομία. Και εδώ θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Σε ποιο βαθμό, γιατί είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται βασανιστήρια και γίνονται μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των αστυνομικών και αστυνομικών που έχουν εκπαιδευτεί από τη UPOL. Και το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό οι δράστες εδώ είναι υπόλογοι έναντι της δικαιοσύνης, προσάγονται στη δικαιοσύνη γιατί νομίζω ότι αυτός θα ήταν ένας ενδεδειγμένος τρόπος να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά ή φαινόμενα στο μέλλον. Επίσης, ε, διατυπώθηκε ε, μια παρατήρηση για τη διαφθορά και θα ήθελα να πω τα εξή. Είναι δύσκολο όταν ε, μιλάμε για διαφθορά στις γραμμές της αστυνομίας και του στρατού αλλά και στους κόλπους της κυβέρνησης. Όταν μιλάμε για διαφθορά εδώ στην κυβέρνηση, ε, τίθε το ερώτημα σε ποιο επίπεδο θα πρέπει εμείς να ε, λειτουργήσουμε. Και όσον αφορά τις εντελώς ε, διαφορετικές αντιλήψεις περί αστυνομίας ή τι τους αντίληψη έχουμε εμείς για μία μη στρατιωτική αστυνομία, υπόθηκε εδώ κατ' επανάληψη ότι οι δικές μας ιδέες επιδέχονται κάποιων διορθώσεων. Η κυρία Γκόμες είπε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να κινηθούμε στην κατεύθυνση μιας ζανταρμερή, μιας χωροφυλακής ενδεχομένω. Εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιη κατά πόσο αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο, στο οποίο θα έπρεπε κανείς να οδηγηθεί. Ο, ο στατηγός ναι είπε ότι υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες και το ερώτημα για μένα είναι, ποιο είναι ποιος είναι ο ρόλος αυτών των παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων στην UPOL ε, και ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία θα έπρεπε να καταλήξουμε εμείς. Κύριε Μπέρκ, αναφερθήκατε σε φαινόμενα πολιτικής ε, ε, διάσπασης. Και αυτό έχει επιπτώσει, το φαινόμενο αυτής της διάσπασης έχει ε, επιπτώσει τη διάσπαση της ίδιας της αστυνομία, του στρατού και των ίδιων των στρατιωτών. Γιατί δεν υπάρχει πλέον καμία συνοχή στους ε, επικεφαλείς του στρατού, οι οποίοι ενδεχομένως θα προτιμήσουν να συνεργαστούν με τους Ταλιμπάν. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το θέμα, πώς το βλέπετε και ποιο μέλλον ε, βλέπετε εδώ με ποιου όρου θα μπορούσατε να το περιγράψετε. Γιατί έχουμε και κάποιε σχετικέ εμπειρίε από το Ιράκ. Πώ ακτιμάτε ε, μετά από 10 χρόνια τη ε, αποστολή τη ε, EU Pol την κατάσταση εκεί ε, δεν ξέρω, αυτό είναι το worst case σενάριο ή υπάρχουν χειρότερα δυνατά σενάρια και αντίστοιχα όπως το Ιράκ ε, υπάρχει εδώ κίνδυνος να ριζοσπαστικοποιηθούν η αστυνομία και ο στρατός στο Αφγανιστάν και να προσρέξουν σε παράνομες πηγές εσόδων και μελλοντικά να υπάρξει ενδεχομένω ένα κενό εξουσίας το οποίο θα έχει επιπτώσεις ε, πολιτικές και θα το εκμεταλλευτούν. Ευχαριστούμε. Μπότιλ Βαλέρο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα βασιστώ και εγώ στη δική μου εμπειρία από πολλά ταξίδια που έχω κάνει στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της εποχής του ISF. Ένα από τα συμπεράσματά μου είναι ότι ε, η εθνική αστυνομία, μια καλώς λειτουργούσα εθνική αστυνομία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση της χώρας και θα πρέπει να μπορούν να την εμπιστεύονται οι πολίτες βέβαια. Από τις επισκέψεις μου αυτές στο Αφγανιστάν είχα θετική εντύπωση από την εργασία εκεί της EUPOL, ε, μόλον ότι ε, πολλά κενά, δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό, δεν μπορούσατε να εξασφαλίσετε το απαραίτητο προσωπικό. Πάντως είχα καλύτερη εντύπωση από την Ιουπόλ από ό,τι είχα από τις υπόλοιπες αποστολές κατάρτισης. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά είχα επίσης την εντύπωση ότι υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν από τις αποστολές αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι καταρτίστηκαν μεν, αλλά κατέληξαν σε άλλες ομάδες μετά, όντας καλύτερα καταρτισμένοι, χωρίς να παραμείνει δηλαδή στην αστυνομική δύναμη του Αφγανιστάν. Θα ήθελα επίσης να είχαμε περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν προχωρήσετε σε κατάρτιση λοιπόν γυναικών αστυνομικών γιατί όσον αφορά τα κοινά εγκλήματα σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά επιτόπου και γυναίκες αστυνομικοί, όσον αφορά την τοπική αυτή αστυνομία, όσον αφορά το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Αναφερθήκατε και στα κίνητρα. Για ποιο λόγο καταρτίζεται κανείς ως αστυνομικός. Είπατε ότι πάρα πολλοί περνούν από προγράμματα κατάρτισης και έπειτα φεύγουν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Να αναφερθώ και σε αυτό που είπε η κυρία Γκόμες πριν από λίγο. Η μεταναστευτική κατάσταση. Ποιε θα είναι οι μελλοντικέ ευρωπαϊκέ δραστηριότητε μετά το 2016. Ξέρουμε ότι έχουμε πλέον μια νέα συμφωνία με το Αφγανιστάν όσον αφορά την μετανάστευση και την επανεισδοχή και γνωρίζουμε επίσης ότι πολλοί μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη είναι από τη φυλή Χαζάρα, όπως είπε η κυρία Γκόμες, Και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ζήσει ποτέ στο Αφγανιστάν, ήταν πάντα πρόσφυγες και ζήσανε σε άλλες χώρες όπως το Ιράν. Και εμείς τώρα ως Ευρωπαίοι τους στέλνουμε σε μια χώρα, το Αφγανιστάν, την οποία δεν την έχουν γνωρίσει μάλλον ποτέ. Είμαι κατά της συμφωνίας αυτής επανεισδοχής. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αποστέλουμε κάποιους ανθρώπους πίσω σε μια χώρα που εξακολουθεί να αποτελεί εμπόλεμη ζώνη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της ε, μετανάστευσης αυτής, τότε θεραπεύουμε απλώς τα συμπτώματα. Θα ήθελα λοιπόν να, μου πείτε τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει επί τόπου. Είναι πλέον έτοιμη η αυγανική αστυνομία. Μπορεί να αναλάβει δράση και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο έργο της αστυνομίας και το έργο των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της εποχής του ISF Ξέρετε ότι ε, την εποχή εκείνη η ΆΕΣΕΦ ασχολείται πάρα πολύ με αστυνομικέ λειτουργίε. Στρατιωτικέ δυνάμει δηλαδή είχαν αναλάβει καθήκοντα αστυνόμευση. Έχουμε καταφέρει να διαχωρίσουμε του δύο αυτού κλάδου. Και ποια πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η μελλοντική πλέον συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Τσέζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχοντας ακούσει τους ε, δύο μιλητές μας, τους οποίους τους άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και πραγματικά τους ευχαριστώ ολόθερμα. Θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε ότι αναδύεται όλο και περισσότερο μία κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Όλο και περισσότερο αποσύρονται οι Ηνωμένε και θεωρώ ότι η απόσυρση αυτή θα επιταχυνθεί μετά την εκλογή του νέου Προέδρου. Υπόθηκε επίσης ότι η σύνθεση των αστυνομικών δυνάμεων θα πρέπει να έχει να κάνει κυρίως με περισσότερους καταρτισμένους πλέον υπαλλήλου, αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε και ποιο ρόλο θα κληθεί να αναλάβει η αστυνομία στο μέλλον. Θα καταφέρει να ξεφύγει από τα στενά στεγανά που έχει αυτή τη στιγμή. Επίσης το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η κοινοτική αποστολή, η ευρωπαϊκή αποστολή στο Αφγανιστάν αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Ιταλοί, χίλιοι περίπου στρατιώτες οι οποίοι έχουν πάει στο Αφγανιστάν και έχοντας έρθει σε επαφή πρόσφατα και με τον πρέσβη της Ιταλίας στο Καμπούλ, γνωρίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο καθότι η αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν είχε πολύ σημαντικό ρόλο με σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι αναγκαστικά απογοητευτικά, γιατί όταν καταρτίζουμε ανθρώπους οι οποίοι στη συνέχεια δεν παραμένουν στην αστυνομική δύναμη της χώρας, τότε αυτό ναι μεν είναι θετικό για την κατάρτιση αυτή καθ' αυτή, αλλά ουσιαστικά δεν συμβάλλει καθόλου σε αστυνομικές δυνάμεις. υπάρχει μια ακτίδα ελπίδας. Κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον καταρτίστηκαν και όχι μόνο τους καταρτήσαμε, αλλά καταφέραμε να τους εμπνεύσουμε, να τους εμφυσίσουμε το κατάλληλο πνεύμα το οποίο πρέπει να έχουν προκειμένου να παραμείνουν σε αστυνομικέ δυνάμεις. Λοιπόν, τον Οκτώβριο είχαμε τη σύνοδο για το Αφγανιστάν και εκεί πέρα δεσμεύτηκαν νέοι πόροι για τη χώρα αυτή. Νομίζω ότι η αποστολή της ΕΟΠΟΛ θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο ή μέχρι τα τέλη του έτους. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η αποστολή αυτή. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να δουμε πως θα συνεχιστει η αποστολη αυτη δηλαδη νομιζω οτι θα πρεπει κατα καποιο τροπο να καταρτίζουμε το προσωπικό της αστυνομίας στο Αφγανιστάν, να συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε τέτοια προγράμματα κατάρτισης. Το προσωπικο της αστυνομια μου λοιπόν είναι το ακόλουθο και απευθύνομαι και στους δύο μιλητές και πραγματικά σε ευχαριστώ. Τι πρέπει ακόμα να κάνουμε τι επιπλέον πρέπει να κάνουμε προκειμένου να καταφέρουμε να συμβάλλουμε πιο αποτελεσματικά και πιο ρεαλιστικά επιτόπου. Ξέρουμε ότι η Ιωπόλ είχε ως στόχο την κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων του Αφγανιστάν. Πώς μπορεί η κατάρτιση αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική και πώς μπορούμε να αποφύγουμε όλα τα αρνητικά τα οποία μας περιγράψατε εσείς σήμερα το πρωί γιατί το είπε και ο επικεφαλής ε, της ε, αντιπροσωπείας για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αφγανιστάν, υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να δαπανούμε ακόμα δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για να αποσυρθούμε κι εμείς όπως οι Αμερικάνοι. Όπως σας είπα εμείς ως Ιταλοί είμαστε επιτόπου και πραγματικά έχουμε συμβάλει πάρα πολύ και έχουμε χάσει μάλιστα και στρατιώτες μας στο Αφγανιστάν. Είμαστε ακόμα παρόντε στο Αφγανιστάν. Θέλουμε να παραμείνουμε στο Αφγανιστάν. Το πιο σημαντικό όμω είναι όλε αυτέ οι αποστολέ, οι οποίε χρηματοδοτούνται άμεσα από την Ευρώπη, να καταλήξουν να γίνουν τελικά λίγο πιο αποτελεσματικέ. Τι μπορούμε να κάνουμε, δώστε μας εσείς ως εμπειρογνώμονες, εμά εμάς ευρωβουλευτές, κάποιες ενδείξεις για το πώς θα μπορούσαν οι αποστολές αυτές να γίνουν κάποιες πιο αποτελεσματικές. Ο κύριος Φρανσούλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια που οργανώσατε αυτήν την ακρόαση. Το αφγανικό είναι παλιό ζήτημα, αλλά θα συνεχίσει να απασχολεί. Από το Μέγα Αλέξανδρο ο πόλεμος. Και κατά όλη την ιστορία της χώρας υπήρχαν σύγκρουσεις συνέχεια. Εισβολές, μάχες, δολοφονίες, βεντέτες κλπ. Mission, European ε, Union with the NATO missions in Afghanistan. Έχουμε τώρα την αποστολή του ΝΑΤΟ. Ο σκοπός είναι να γίνει κάποιο είδους ανασυγκρότηση της χώρας. Να καταστεί το κράτος βιώσιμο και να αποκτήσει την ενότητα που ουδέποτε είχε. Ουδέποτε υπήρξε ενότητα στη χώρα. Όπως γνωρίζετε. Ήταν πάντα οδυνηρή η ιστορία της χώρας και αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διαμεσολαβήσει, να παράσχει ε, συμβουλές στους εμπλεκομένους και στους ενδιαφερόμενους. Μιλώ και για τους γείτονες της χώρας. Κίνα, κυρίως το Πακιστάν, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Κυργιστάν, επίσης ε, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα Θα πρέπει δύο προς το χρόνο να συναντώνται όλοι αυτοί και να συζητούν το πώς έχει κατάσταση στη χώρα, ούτω ώστε να βρεθεί ένα κοινό τόπος, γιατί όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά τα ξένα συμφέροντα. Δυστυχώς. Και την ύφη την πληρώνει για αυτά τα ξένα συμφέροντα ο λαός. Και ξέρετε ποια είναι η πηγή του κακού. Και αυτό έχει σχέση με το ρόλο της Ένωσης. Το 1995. Η συνολική γραμμή που χαράχτηκε μεταξύ Αφγανιστάν και της πρώην Βρετανικής Ινδίας. Όμως το, τα σύνορα με το Πακιστάν τώρα δεν γνωρίζονται ούτε από την άλλη χώρα. Να, ποιο είναι το βασικό καθήκον της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Να κλειστεί μια συμφωνία μεταξύ των χωρών για να αναγνωριστούν τα σύνορα. Και το 1795 όταν χάριξε τα σύνορα τότε ο Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, τι έκανε. Άφησε 15-16 εκατομμύρια παστούν στο Αφγανιστάν και άλλα 20 εκατομμύρια στο Πακιστάν και να η βασική αιτία των προστριβών των Παστούν μεταξύ των, των Τατζίκων που είναι 29% των Χαζάρων, των Μογγόλων που αναφέρατε, των ε, που είναι κοντά με το Ιράν και, και των άλλων ε, Βαλούχων, Βελούχων κλπ. των άλλων φυλών των άλλων ε, εθνοτικών μειοτήτων στη χώρα. αυτά τα σαφή σύνορα που υπάρχουν και κόβουν τη χώρα στα δύο μεταξύ βορρά και νότου τα θεωρητικά σύνορα. Συμπαθείτε με, αλλά έχω γράψει ένα βιβλίο το 2013, συγγνώμη που σα το λέω, όσον αφορά την ε, περίπλοκη αυτή εξίσωση που λέγεται Αφγανιστάν. Είναι μια εξίσωση που κανείς δεν κατάφερε να λύσει. Και θα εκρεμεί άλυτη αυτή η εξίσωση. Για πάντα εάν δεν εξετάσουμε τις πραγματικές ρίζες του προβλήματος. Και πάλι σας ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις σας, αλλά εάν δεν υπάρξει συνεννόηση των γειτόνων και των μεγάλων δυνάμεων, δεν πρόκειται ποτέ να ανασυρωτηθεί η χώρα, να γνωρίσει την ενότητα και την ειρήνη. Ακριβώς γιατί εκεί πέρα έχουν πέσει τόσα πολλά μεγάλα ισχυρά συμφέροντα. Ευχαριστούμε κύριε Φροντζουλίγα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πραγματικά εντυπωσιακέ σας παρατηρήσεις. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών, αλλά θα ήθελα να θέσω κι εγώ μια ερώτηση προς τους δύο ομιλητές, κυρίως όμως τον κύριο Μπέρκερ αναφέρατε τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τα διαφορετικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν εντός της eu Ότι υπάρχουν ε, κάποιοι που έχουν μια εμπειρία στο, στην ε, γαλλική ζωνταρμερή, στη χωροφυλακή. Υπάρχει αυτό το μοντέλο της γαλλικής, γαλλικής χωροφυλακής ε, και ενδεχομένως υπάρχουν κάποια άλλα μοντέλα, το βρετανικό κλπ. Ε, ποιο μοντέλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ισχύσει για την κατάρτιση στο Αφγανιστάν αλλά και για τις ε, παρατηρήσεις της, της κυρίας Ανζελίκας. Αναφερθήκατε δεύτερον ε, σε μια διαφορά προτεραιοτήτων μεταξύ της EU Pol ή του βασικού της πυρήνα από τη μία και των ε, Καναδών και των, και των Ορβηγών. Θα μπορούσατε παρακαλώ να πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα και το τρίτο μου ερώτημα αφορά το εξής. Αναφερθήκατε στην επίσημη και ανεπίσημη ε, ύπαρξη ισχύ του Ισλαμικού νόμου. Ποια είναι η δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ αστυνομίας ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, ε, έρευνας και ανάκρισης και των παραδοσιακών ε, μορφών. Τι εκπαίδευση, ποιο μοντέλο εκπαίδευση θα έπρεπε να ισχύσει εδώ, ούτως ώστε να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Γιατί υπάρχουν πολλές ανησυχίες συναδέλφους, τις συμμερίζομαι και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, προσπάθειές σας. Και πραγματικά θα θέλαμε να αποτίσουμε τιμή ε, σε όλους όσους ε, πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν και να προσπαθούν για ένα καλύτερο μέλλον στο Αφγανιστάν, όλα τα μέλη των Αποστολών. Έχετε το λόγο ο κύριος Βέρσμανς καταρχήν και ο κύριος Μπέρκ ε, στη συνέχεια. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Εγώ μπορώ να απαντήσω κυρίως σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν ε, με την EU Poll, γιατί αυτή είναι η βασική μαρμοδιότητα και απαντώντας βέβαια σε ερωτήσεις αυτές, θα πρέπει να συνδέσω τις απαντήσεις αυτές με την ίδια την εντολή της EUPOL. Για παράδειγμα, η EUPOL δεν συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία του Αφγανιστάν. Έχουμε ασχοληθεί κυρίως με την εθνική, κεντρική δηλαδή αστυνομία του Αφγανιστάν. Τα βασικότερα στοιχεία από τη συζήτηση αυτή, όπως προκύπτουν και από αυτά που, είπε η κυρία Γκόμες, είναι το τι συνέβη αρχικά με το προσωπικό το οποίο στελέχωνε το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς επίσης και το δικαστικό σύστημα της χώρας. Υπήρχαν εκεί πέρα αρκετά κενά και το όλο περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο στο Αφγανιστάν. Όσον αφορά καταρχάς την κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτό το οποίο έχει προκύψει από την συζήτηση είναι ότι η πρωταρχική θέση έχει η πολιτική Και σε αυτό εντάσσω βέβαια και την κοινοβουλευτική εξουσία, την κοινοβουλευτική διάσταση. Προφανώς λοιπόν ήμασταν σε επαφές με τους, κοινοβου... με τους βουλευτές στο Αφγανιστάν και μας ενδιέφερε και εμάς ιδιαίτερα να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην αστυνομία. Τώρα, το αν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε όλο και περισσότερο με τις ήδη φυστάμενες δυνάμεις, Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι μια τέτοια συνεργασία θα λειτουργούσε σωστά και επί τόπου, ότι θα ήταν δηλαδή θετική και από επιχειρησιακής πλευράς. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα. Αξιολόγηση τώρα των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω μόνο για το Υπουργείο Εσωτερικών, για κανένα άλλο θεσμικό όργανο. Και όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, Είδαμε να σημειώνεται πρόοδο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά υπάρχουν επίσης και κάποια δύναμα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω πάντως ότι ε, η, αστυνομία, ε, η αστυνομική αυτή αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε να συμβάλλει στην θετική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και στη δημιουργία ενός καλύτερου συστήματος συντονισμού των δραστηριοτήτων του. Η ίδιο πόλοντο είδε μία αλλαγή στην εντολή της, αυτό αληθεύει. Χρειάστηκε να προσαρμόσουμε την εντολή γιατί συνεχώς κάνουμε αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις των όσων συμβαίνουν επί Ξέρετε ότι όταν ξεκινάει μία αποστολή Πάντα υπάρχουν διδάγματα τα οποία αντλούνται κατά τη διάρκεια της αποστολής, δεν είναι ποτέ δυνατόν εκ των προτέρων να γνωρίζουμε τα πάντα. Γίνονται λοιπόν ανατακτικά χρονικά διαστήματα αναθεωρήσεις, επικαιροποίησει και προσαρμόζουμε κάθε φορά μία αποστολή στις επιτόπου ανάγκες και προσδοκίες. Αντλούμε δηλαδή διδάγματα από την επιτόπου κατάσταση. Σαφώς θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα όσα ισχύουν επιτόπου και γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει να έχουμε και ισχυρά προγράμματα κατάρτισης είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε καλά καταρτισμένους υπαλλήλους. Τα όσα άκουσα ως προβλήματα θεωρώ ότι είναι αρκετά μεμονωμένα. Η αστυνόμευση και οι υπηρεσίες αστυνομίες είναι όλο και πιο απαραίτητες για το Αφγανιστάν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολιτική μη στρατιωτική αστυνομία ή ακόμα και για τοπική κοινοτική αστυνόμευση, για το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Η προσέγγιση όμως που αναφέρατε εσείς της ζωνταγμερή, της χωροφυλακής, είναι μια προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει άλλοι διεθνείς φορείς επιτόπου. Εμείς επικεντρωθήκαμε κυρίως σε ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά σε μία περίοδο μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης στην οποία βρισκόμαστε και γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να θέσουμε εμεί τα θεμέλια για μία μη στρατιωτική αστυνομία η οποία θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε καθήκοντα όπως εγκληματικές έρευνες, αστυνόμευση βάση βιστευτικών πληροφοριών και το καθεξής. Η συμμετοχή τώρα των γυναικών σε αστυνομικέ δυνάμεις και αυτό αποτέλεσε έναν από τους στόχους μας. Έχουμε ε, θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να συμπεριλάβουμε περισσότερες γυναίκες. Είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και τα κατάλληλα συμβούλια στην οποία, στα οποία θα συμμετέχουν οι γυναίκες αστυνομικοί. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε όλα αυτά τεχνικές διευθετήσεις τελικά στα πλαίσια ενός γενικότερου περιβάλλοντος που παρουσιάζει πάρα πολλές προκλήσεις. Όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, εμείς ως αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν και κινούμενοι στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της μετανάστευσης. Αλλά στα πλαίσια των εγκληματολογικών ερευνών, των ποινικών ερευνών, προφανώς ασχοληθήκαμε και με την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων διακίνηση μεταναστών. Όσον αφορά τώρα τη χρησιμοποίηση βασανιστήριων, έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πέρα ένα συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, προσπαθώντας να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα χρησιμοποίησης βασανιστήριων. Τονίστηκε επίσης η περιφερειακή διάσταση. Νομίζω ότι αυτή υπερβαίνει όμως την αποστολή της Ιγιουπόλ. Έχουμε όμως έναν ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με την περιφερειακή διάσταση και ο οποίος ήταν και παρόν στην διάσκεψη που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ για τα όσα ενδιαφέροντα σχολιάσατε. Πρώτα για το Κοινοβούλιο πάντοτε θα πρέπει ε, σε μια δημοκρατία που υπάρχει πολιτικό έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στον προπολογισμό δημοσιότητα των εκταμιεύσεων κλπ. Όμω είπαμε και εκεί πέρα τα τοπικά συμφέροντα που ότι υπάρχει μικροπολιτική ο σεκταρισμό τέλο πάντων και έχουμε, και την αντικατάσταση των αξιωματούχων ανάλογα με τα συμφέροντα. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε όλη αυτή την ε, ε, ανεπιθύμητη παρέμβαση στο έργο τη Και Το που δεν συμβαδίζει με το αν θέλουμε να χτίσουμε καλή διοίκηση. Και όσον αφορά τώρα τη δική μας οργάνωση, βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση, αναθεώρηση τη ε, ιστορικής μας, της, πολιτικής μας άμυνας. Να υπάρχει ένα πρότυπο εκπαίδευση αστυνομία από πλευρά Ευρώπη. Θα πρέπει να στοχεύεται κάθε χώρα. Θα πρέπει να ξέρουν γλώσσε οι αστυνομικοί, να ξέρουν το δίκαιο της χώρας εκεί όπου θα αποσπαστούν. θα βοηθούσε να ήξερα να πούμε τον Ισλαμικό νόμο να μπορούσαν να συνοηθούν με τη διοίκηση. Δεν μπορεί ο, να βγαίνει και ο Άγγλος και να μιλάει με το αγγλικό πρότυπο και ο Γάλλος ε, να, πώς να με τους τοπικούς με βάση το δικό τους. Έτσι θα πρέπει να δρά μια αστυνομία. Και θα πρέπει να υπάρχει επομένω μια μακρά κατάρτιση αυτών που στέλνουμε εκεί. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους αστυνομικούς και για τους σύμβουλους. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να θέλουν να ένα μοντέλο σε μια ξένη χώρα που δεν είναι εφαρμόσιμο. Έτσι θα πρέπει να ενεργήσουμε στα πλαίσια της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Επίσης, όσον αφορά την αστυνομία της γειτονιάς, θα πρέπει αυτό να γίνει ψηλότερη προτεραιότητα που δεν είναι. Α, άλλο ένα επεισόδιο. Το 11 είχαμε κάποια σύλληψη κάποιου αστυνομικού, δεν το ήξερε αυτό ο μέντορ, πως λέμε, αυτού και είχε συλληφθεί για λόγους διαφθοράς. Όμως ήταν αλήθεια αυτό ή συνελήφθη γιατί είχε ενοχλήσει κάποια συμφέροντα. Δεν ξέραμε. Άρα χρειάζεται να υπάρχει και υπηρεσία πληροφοριών και γνώση των πολιτικών της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να υπάρξει κάποια αποστολή. Και επίσης οι τεχνικές δυνατότητες εκπαίδευσης. Και χρειάζονται όλα αυτά ταυτοχρόνως να συνεπάρχουν. Επίσης, ε, το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει κάποιες ειδικές δυνάμεις αστυνομία. και Δυστυχώ, ανάλογα με τις ε, επιδόσεις ή τα αποτέλεσματα κάθε προσπάθειας ε, υπήρχε επικάλυψη, υπήρχε επανάληψη αυτής της προσπάθειας και φτιάχνανε καινούργια ε, τέτοια η ειδική, η ειδική επαναληψη αυτή της προσπάθεια και φτιαχνανε καινουργια τετοια η ειδικη ειδικη δυναμη της αστυνομία καθε χρονο Η ιδεολογία επίσης επηρεάζει το έργο του Υπουργείου των Εσωτερικών και έτσι υπάρχουν προσπάθειες ελέγχου του έργου των εισαγγελίων και όχι μόνο. Θα πρέπει κανείς να καταλάβει αυτές όλες τις δυναμικές. Αλλά βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και υπηρεσία πληροφοριών που να βοηθά. Έχουμε την ανκόπια και τις ειδικές δυνάμεις αστυνομίας. Αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο τι αρμοδιότητες έχει η κάθε υπηρεσία. Υπήρχαν κεντροκατευθυνόμενες τάσεις και ε, αποκεντρωτικές, ας πούμε. Αυτά δεν είχαν ξεκαθαριστεί που θα πρέπει αυτό να γίνει. Δεν εκπαιδεύσαμε τους ΑΝΚΟΠ, αλλά είχαμε πολλούς ε, χωροφύλακες, ζεντάρμ μαζί. Δεν έκαναν αυτή καμία εκπαίδευση. Και τελικά θα έπρεπε να προσέξουμε ποιοι από τους αστυνομικούς που είχαν μαζί μας από την Ευρώπη είχαν γνώσεις που τέριαζαν με το σώμα το οποίο εκπαίδευαν. Τώρα, τι γίνεται με τους ε, Χαζάρους. Είχαμε τον αντιπρόεδρο Χαλίλη. Και Τώρα οι Χαζάρι θέλουν να αντιδράσουν, ετοιμάζονται για αντιπαράθεση. Είναι η μόνη ομάδα που είχε αφοπλιστεί με τη συμφωνία TDR. Τους πληρώσαμε για να καταθέσουν τα όπλα, αλλά τώρα ξαναμαζεύουν όπλα. Όντως είναι πάντως σε ευάλωτη θέση και κάποιος θα τους υπερασπιστεί. Τώρα όσον αφορά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά ε, τις καταχρήσεις. Οι Καναδοί ε, προσπάθησαν να αλλάξουν την κατάσταση, θεωρούσαν ότι υπήρχαν ε, βασανιστήρια και δεν θέλαν να δώσουν στις αφγανικές αρχές κάποιους φυλακισμένους. Η NDS ήταν ευχαριστημένοι που είχαν πάρει αυξημένες αρμοδιότητες, αλλά τι μας χρησιμοποιούσαν, μήπως. Να, ας πούμε, ήταν αυτό ένα επεισόδιο όπου η Γιούπολ παγιδεύτηκε. Πρέπει να προσέξουμε, επομένως, να μην παρασυρώμαστε από κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι θετικό. Όχι, πρέπει να προσέχουμε και πάντοτε η αρρωγή μας να έχει ως προϋπόθεση τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να γίνουν. DNP και DNA δρούν χωρίς συνέπεια μεταξύ της δράσης της μιας περισσίας και την άλλη. Είπαμε ότι το ΝΑΤΟ έκανε ό,τι ήθελε, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε ενιαία δράση. Επομένως, αυτή η έλλειψη συνοχής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ στρατού και αστυνομία στο Αφγανιστάν. Άρα και αυτά θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να τα λάβουν υπόψη. Για το Ισλαμικό Δίκαιο, τον Ισλαμικό νόμο τώρα, προηγουμένως στο Αφγανιστάν υπήρχε μετριοπαθής εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Παλιότερα οι δικαστές πηγαίνουν στο Κάιρο, τώρα πάνε στο Πακιστάν, όπου εκεί είναι πιο ριζοσπαστικό, πιο αυστηρό το Ισλαμικό δίκαιο. Εμείς δεν θα πρέπει να προσπαθούμε μόνο να εξάγουμε τα δικά μας μοντέλα, το δικό μας δίκαιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ρόλο του Ισλαμικού νόμου στη χώρα και να ασχοληθούμε να δούμε τι είδου Ισλαμικό νόμο θέλουμε, τι από όσα γίνονται συνάδουν προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περισσότερο να ασχοληθούμε με τον Ισλαμικό νόμο και όχι μόνο με τα κοσμικά όπως έχουν δίκαια. Αυτό θέλει ο λαός του Αφγανιστάν. Και η αστυνομία λέει ότι η Ταλιμπάν είναι ηθικός παραγόν. Αυτά όταν δεν πολεμά η αστυνομία με ναι, τους Ταλιμπάν. Οπότε δεν είναι κακό αυτό. Να μην το βλέπουμε, τους, το, το, βλέπουμε σαν μαύρο άσπρο. Γιατί σε κάθε μέρος η κατάσταση είναι διαφορετική. Αλλάζουν πλευρά πολύ, ανάλογα με το αν έχουν εξουσία κλπ. Φυσικά και δεν μπορούμε να δεχθούμε όλους τους στόχους των ε, Ταλιμπάν που λεμάνε όλη την ώρα, αλλά σε κάποιες επαρχίες είναι μέρος του κατεστημένου, ας πούμε. Αλλά φυσικά και ενώ άλλο αστυνομία, άλλο Ταλιμπάν πολλές φορές μπορούν να δράσουν από κοινού, να συνοηθούν τοπικά. Υπάρχουν πολλέ οργανώσει που δρούν εκεί, κάνουν για αξιολόγηση. Και στην, ε, στην Ιρλανδία τώρα έχουμε ένα ίδρυμα που έχει δημοσιοποιήσει κάποιες πολύ αξιολόγες εκθέσεις. Αν θέλουμε επομένω να συζητήσουμε στα σοβαρά με τους Αυγανού εταίρους, θα πρέπει να βάλουμε κάποιες προϋποθέσεις στις σχέσεις μας, στη βοήθειά μας. Προστασία των υπηρεσιών της χώρας, να ρωτήσουμε διαφάνεια. Και αφού μιλούμε για επαναπατρισμό των ετούντων άσυλο, αυτό το ξέρουν. θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή μας τη θέση, γιατί Αυτά έχουν σημασία για εκείνους. Άρα και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι όρος και προϋπόθηκε για την περαιτέρω συνεργασία. Εύκολο να λες ότι είσαι φίλος και ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά τελικά θα πρέπει κανείς να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι όταν διακυβεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και τιμίο δεν σημαίνει ότι αν θέλουμε το καλό της χώρας θα πρέπει να λέμε ναι σε όλα να είμαστε συγκαταβατικοί. Thanks a lot. Uh, Burke... Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρκ. Θα ήθελα να διευκρινίσω την ερώτησή μου γιατί δεν αφορούσε τον Ισλαμικό νόμο. Το αναγνωρίζω ε, δεν το θέτω να αμφιβόλω. Ήταν απλώς μια περιέργεια εκ μέρους μας. Κατά πόσο μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της αστυνομίας την οποία εκπαιδεύουμε, δηλαδή του ευρωπαϊκού μοντέλου της αστυνόμευσης και της δικαστικής εξουσίας η οποία λαμβάνει υπόψη στην Ισλαμική νομολογία. Αυτή η δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ των δύο. Παρακαλώ. Και κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να αναφερθεί τις καναδικές και νορβηγικές ε, προτεραιότητες. Ναι, ε, ρωτάτε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Αστυνομεύση... Ενδεχομένως δεν κατάλαβα και πάλι την ερώτησή σας, ε, λέει ο κύριος Μπέρκ. As Όπως αναφέρατε ορθά, ε, υπάρχει Ισλαμική νομολογία στο σύστημα δικαιοσύνης του Αφγανιστάν. Θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τη δική σας γνώμη εν σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ανακριτικές ε, αρμοδιότητες που μπορεί να έχει η αστυνομία και κατά πόσο μπορούν να διαχωριστούν από το σύστημα της δικαιοσύνης. Το άλλο θέμα αφορούσε την και την, τον Καναδά και την Νορβηγία. Ε, ναι, ανησυχώ, ε, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν είναι ξεκάθαρος αυτός ο διαχωρισμός και διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Ε, και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες επικάλυψης ε, και ορισμένες φορές υπάρχει και αντίφαση ε, όσον αφορά τον ε, νόμο περί αστυνομίας, όπου υπάρχουν διάφοροι σύμβουλοι οι οποίοι πιέζουν ε, σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ οι Αφγανοί εταίροι προσπαθούν επίσης να ευχαριστήσουν διάφορα υπουργεία. Όσον αφορά την, το τμήμα πάταξης του εγκλήματος, αυτοί βλέπουν το ρόλο τους πολύ διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την EU Υπάρχουν εξαιρετικοί μέντορες της EUPOL οι οποίοι προσπαθούν να κατατήσουν κάποιο άτομα που θα ακριβώς θα λειτουργούν ως συνδετική κρίκη μεταξύ αστυνομία και δικαστικών οργάνων. Όπως σας είπα υπάρχουν αντιφατικοί μεταξύ τους κώδικες και νόμοι. Ε, συμφωνώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό έλλειμμα γιατί μιλάμε για... Ε, ε, γιατί ο ρόλος του ΝΑΤΟ, οι εκλογές, όλα αυτά μας αποσπούν από τα ουσιαστικά προβλήματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Ε, θεωρώ, όπως σας είπα, ότι ποικίλει ανάλογα με την περιοχή έχουμε πολύ καλούς αξιωματούχους της αστυνομίας οι οποίοι οποίοι μπορούν να συντάξουν πολύ καλές εκθέσεις, να τις διαβιβάσουν στη συνέχεια στην εισαγγελία κλπ. Αλλά η κατάσταση αυτή πραγματικά είναι απογοητευτική. Για τους μέντορες υπάρχουν ε, θεμελιώδη θέματα όσον, αφορούν, όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν σημαντικά και για μας και για τους Ευρωπαίους ε, αξιωματούχους πραγματικά είναι σημαντικό το σχόλιά σας. Τώρα όσον αφορά τον Καναδά και την Ορβηγία ή ε, ε, τη Νέα Ζηλανδία, εγώ χρησιμοποίησα αυτές τις χώρες σαν παραδείγματα τα οποία ήταν υπό την αιγίδα της UPOL. Ε, αλλά πραγματικά δέχονται πιέσεις από τις δικές τους κυβερνήσεις εν σχέση με τις ομάδες αναποκατάστασης της χώρας. Και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τελικά ε, πληρώνουν για αυτές τις αποστολές ε, για να κάνουν το έργο τους. Και υπάρχουν, όπως σας είπα, άλλα συμφέροντα. Υπάρχει ομάδα ε, αποκατάστασης της, που προσπαθεί να αναδομήσει τη χώρα και η οποία έχει άλλα συμφέροντα και ακολουθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Ε, καμιά φορά ε, όταν υπάρχει μια τεράστια αποστολή του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ ε, είναι πολύ δύσκολο να λάβουν υπόψη τους τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ενώ εμείς ε, χρηματοδοτούμε τις ε, δικές μας αποστολές βασιζόμενοι σε ένα εντελώ διαφορετικό πρόγραμμα. Ελπίζω ότι εν μέρει να απάντησα το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η μερίσια διάταξη για την πρωινή μας συνεδρίαση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις που κάνανε, για το ότι απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Προφανώς θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το Αφγανιστάν Καταλαβαίνετε το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δεν πρόκειται να περιορίσουμε την εξέταση στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και εσείς είστε επίσης παρόντες στις 3 το μεσημέρι για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ.